Τα συνοπτικά πρακτικά της 25ης ε, Δευτέρου έχουν διανεμηθεί. Δεν έχετε αντιρρήσει από ό,τι βλέπω. Κυρίες και κύριοι, εξ ονόματος του Αντιπροέδρου κυρίου Ταγιάννη θα ήθελα να σας ενημερώσω για κάτι που με παρακάλεσε. Έξω από την αίθουσα της Ολομέλειας θα βρείτε φυλάδια που έχουν εκπονήσει υπηρεσίες σε συνεργασία με τον κύριο Ταγιάννη και αφορούν ε, τα θέματα ασφαλείας και τους κανόνες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και παρακαλείστε να ενημερωθείτε. Ο κύριος